Please leave the room. Παρακαλώ πολύ ησύχω να εγκαταλείψετε την αίθουσα. Because itre to start a boat. Yeah. Fuori. Λοιπόν, ε, λοιπόν. τις εργασίες της Επιτροπής Ήτρε. Γνωρίζετε ότι θα αντιμετωπίσω με κάποια προβληματάκια διότι δυστυχώς έχουμε βεβαρημένη ημερήσια διάταξη με πολύ λίγο χρόνο αλλά όλα αυτά που είχαμε εγγράψει στη μέση διάταξη είναι υποχρεωτικά γιατί υπάρχουν χρονικά περιθώρια τα οποία πρέπει να σεβαστούμε. Θα πρέπει επομένως να προσπαθήσουμε να μειώσουμε στο ελάχιστο, στο ελάχιστο λέω, και τον χρόνο εργασίας και τον χρόνο παρεμβάσεων. Μου ζητήθηκε να περιμένω ακόμα ένα λεπτάκι έτσι ώστε να ηρεμήσει η αίθουσα οι συνάδελφοι που έφυγαν για λίγο και εγκατέλειψαν την αίθουσα να ξανά πάρουν τις θέσεις τους. Θα διακόψουμε λοιπόν και μετά από ένα λεπτό θα ξαναρχίσουμε με την ψηφοφορία. Ξέρετε ότι έχουμε δύο ψηφοφορίες που πρέπει να γίνουν πολύ γρήγορα, αλλά μετά έχουμε και ένα πρόβλημα. Δηλαδή έχουμε μία σειρά ζητημάτων και ε, ε ε, επί των οποίων έχουμε μεγάλη καθυστέρηση. Να ξαναρχίσουμε λοιπόν, ρωτάει η Πρόεδρος, να ξαναρχίσουμε. Πρώτα απ' όλα, να κάνουμε μία ενδεικτική ψηφοφορία έτσι ώστε ε, να δούμε ότι μπορούν να ψηφίσουν όσοι έχουν δικαίωμα ψήφου Γι' αυτό λοιπόν να κάνουμε μια ε, δοκιμαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Ε, proviamo a verificare i presenti, prego. Μια υπαλήθευση παρουσιών λοιπόν. Παρακαλώ. Bene. E λοιπόν, τα καταφέραμε από ό,τι φαίνεται. Υπάρχουν ε, όσε ψήφοι πρέπει να υπάρχουν, άρα μπορούμε να ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία ε, της εκθέσεως Ulfskog. Ξεκινάμε λοιπόν με μία ψηφοφορία en bloc από την τροπολογία 33 μέχρι την 48. Με παρακολουθείτε όλοι. 33 μέχρι 48 υπέρ. Κατά. Νομίζω πως εγκρίνονται, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε αυτή την ηλεκτρονική επαλήθευση. Παρακαλώ. Ψηφίζουμε λοιπόν από την τροπολογία 33 μέχρι την 58 λέει η Πρόεδρος. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας. 20 ψήφοι υπέρ, 17 κατά, επομένως εγκρίνεται. Περνάμε τώρα σε μια δεύτερη σειρά ε, τροπολογιών από την 34 μέχρι την 26. Όχι, κάνω λάθος. Όχι, έτσι είναι. 34, 41, 42, 25, 26 υπέρ. Κατά απορρίπτονται. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 35. 35 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 36 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. Τροπολογία 37 <clears throat> υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση από τις τροπολογίες 7 παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 14 ψήφοι υπέρ, 26 κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 40, δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ο μπλοκ. την 8, την 17, την 19, την 18, την 20 και την 5. Μέχρι την 5 λοιπόν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση επί του συνόλου αυτών των ε, ψηφοφοριών, πολύ ωραία, των τροπολογιών, συγγνώμη, άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογίες 8 ε, μέχρι 5 πέρας της ψηφοφορίας. 16 ψήφοι υπέρ, 24 κατά, επομένως απορρίπτονται. Τροπολογία 75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογίες από 9 μέχρι 16 on block. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 43 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 44 ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 43 παρακαλώ άρχεται η ψηφοφορία πέρας 22 υπέρ 16 κατά ζητώ συγγνώμη όντως ενεκρίθη τροπολογία 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται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 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60-61 μαζί υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 62, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 63, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 64 και τροπολογία 65 από κοινού, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Τροπολογία 68 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 και τροπολογία 6 δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 30 υπέρ. Κατά η ηλεκτρονική επαλήθευση από της τροπολογίας 30. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία λοιπόν επί της τροπολογίας 30 πέρας της ψηφοφορίας 15 υπέρ 25 κατά απερίφθη. Τροπολογία 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 69, 70 και 31 από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 71, τροπολογία 72 και 32 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Νοντε. Τροπολογία 74 υπέρ κατά 74. 74. Τροπολογία 7-4, 74, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 77, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 1, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 23 υπέρ. Ο, ηλεκτρονική επαλήθευση από τις τροπολογίες 22. Παρακαλώ, ηλεκτρονική ψηφοφορία λοιπόν. Τροπολογία 22. Πέρας της ψηφοφορίας απερίφθη. Τροπολογία 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Παρακαλώ, άρχεται. Πέρας. 24 ψήφοι υπέρ, 14 ψήφοι κατά μία αποχή ε, εγκρίνεται και συγχαίρουμε την εισηγήτρια. Περνάμε τώρα στην επόμενη ψηφοφορία. Είναι η ψηφοφορία της εκθέσεως Βαλεάν.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 αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 40 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Τροπολογία 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Τροπολογία 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 47 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 6 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 48, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 52, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 53, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 54, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 17, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 55 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 18 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 56 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 19 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 57 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 58 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 59 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 60 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμό 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 24 υπέρ κατά αποχές. Συγγνώμη, έκανα κάποιο λάθος. Τροπολογία 24, υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 25, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 1, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία η ηλεκτρονική επαλήθευση επί της τροπολογίας 2 βεβαίως άρχεται η ψηφοφορία. Επί της τροπολογίας 2 πέρας της ψηφοφορίας. 11 ψήφοι υπέρ, 30 ψήφοι κατά, ζητώ συγγνώμη, απερίφθη. Τροπολογία 27 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 28 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, συμβιβασμός 3 υπέρ κα... Συμβιβασμός 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 36 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παρακαλώ. θα δεχθώ το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας γιατί αυτή είναι η δουλειά μας, αλλά δεν είναι καλή ιδέα μετά από τόσο έντονες ψηφοφορίες να ξαναψηφίζουμε. Γιατί βλέπετε ότι είμαστε πάρα πολύ λίγοι και αυτό δεν είναι καθόλου σωστό. Νομίζω λοιπόν ότι θα έπρεπε να ψηφίσουμε μόνο το μεγάλο, το κύριο θέμα το πρωί και τίποτα άλλο μετά. Ευχαριστώ ε, τον Κλόντο για αυτό το οποίο είπε και για τις ανησυχίες τις οποίες εξέφρασε αυτός και οι συναδελφοί του για τις διαδικασίες. Το πρόβλημά μου δεν ήταν αυτό εμένα. Το πρόβλημά μου είναι ότι όλες αυτές οι τροπολογίες μας έφτασαν πάρα πολύ αργά. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε δεν είναι καθόλου ε, καλή. Δεν μας τιμά αυτό το οποίο έχει γίνει και θα επανέλθουμε ελπίζω. εγώ ε, λέει ο μιλητής ε, δεν κατανοώ αυτά τα οποία είπε ο κύριος Τούρμες. Μιλάμε αυτή τη στιγμή για νομοθετικές ρυθμίσεις που μπορεί κύριε Τούρμες να ζώσουν πάρα πολλές ζωές στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα χρόνια. Ίσως το θέμα αυτό να είναι πιο σημαντικό από το προηγούμενο. Κοιτάξτε, ευχαριστώ τον κύριο Τούρμες για τις παρατηρήσεις του. Έτσι και αλλιώ θα έχουμε την τελική ψηφοφορία και στην άλλη αρμόδια επιτροπή στις 24 Ιανουαρίου. Κοιτάξτε, ίσως με παρανοήσατε. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι σημαντική η ψηφοφορία. Θα αναγνωρίζαμε τη σημασία της όμως αν την ψηφίζαμε μόνη της. Ξέρω ότι έτσι κι αλλιώς έχουμε πρόβλημα χρόνου, λέει ο κύριος Τούρμες, δεν θα επιμείνω. Κοιτάξτε, φτάνουμε στην τελική ψηφοφορία. Λοιπόν, ψηφίζετε. Τέλος της ψηφοφορία. 34 υπέρ, 4 κατά, 3 αποχές. Γίνεται δεκτή. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους λοιπόν για την παρουσία τους εδώ. Περνάμε στο επόμενο θέμα, το οποίο είναι και αυτό απαραίτητο. Καλά θα ήταν να φεύγαμε όλοι, αλλά έχουμε το σημείο 6 στην ημερήσια διάταξη. Έχουμε το θέμα που αφορά το λεγόμενο πακέτο καινοτομίας τον ορίζοντα 2020 και την απαλλαγή. Ε, ε, Έχουν φύγει πάρα πολλοί συνάδελφοι, αλλά εδώ υπάρχουν ορισμένοι συνάδελφοι και θα τους δώσω το λόγο. Θα ξεκινήσω με τον κύριο Έλλερ. Κυρίες και κύριοι, την περίπτωση αυτή δεν μιλώ εξ ονοματός μου, αλλά η κυρία Γκρέσλε με παρακάλεσε για λογαριασμό των συναδέλφων της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού να αναγνώσω μια σύντομη δήλωση για τα θέματα. Δυστυχώς υπάρχουν άλλα ανοιχτά μικρόφωνα και ο Διερμιάς δεν καταλαβαίνει καλά. Πρόκειται για τα joint undertaking. Γνωρίζετε ότι όλες οι πολιτικές ομάδες έχουν καταθέσει διαφορετικές ρυθμίσεις για τις απαλλαγές. Μαζί με τους συναδέλφους των Επιτροπών Προϋπολογισμών και Ελέγχου του Προϋπολογισμού και επιθυμώ, λέει η κυρία Γκρέσλε, να ευχαριστήσω τα δύο άλλα θεσμικά όργανα, Συμβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι έχουν γίνει προηγουμένως συνομιλίες με κατεύθυνση μια συμφωνία που να μπορέσει να στηριχθεί από την πλειοψηφία των πολιτικών ομάδων. Η κυρία Γκρέσλε λοιπόν λέει όπως θα μπορέσουν να επιβιώσουν και εκπρόσωποι του Συμβουλίου η Κορεπέρ χθε δέχθηκε την κοινή δήλωση με την οποία τα τρία θεσμικά όργανα συμφωνούν επί διαδικασίας. Η περαιτέρω διαδικασία στο Κοινοβούλιο θα έχει ως εξής. Στην βάση της διαβεβαιώσεως που δίνει το Συμβούλιο, ο συντονισμός οι συντονιστέ, μάλλον των Επιτροπών Προϋπολογισμών και Ελέγχου Προϋπολογισμού θα προχωρήσουν σε κοινή δήλωση για το ψήφισμα, θα αποσύρουν δηλαδή το ψήφισμα ενστάσεως κατά των ε, πράξεων. Στην Ολομέλεια θα λάβουν τον λόγο ο κύριος Λαμασούρ και ο κύριος Κόνραντ για να αναγνώσουν σύνοψη της κοινή δηλώσεως και να αποσύρουν στο όνομα των συντονιστών το ψήφισμα. Θα δώσει δε τελική μορφή το Συμβούλιο και από το Κοινοβούλιο θα δοθεί τελική μορφή πριν από την συνέχιση διαδικασίας. Ευχαριστώ, λέει κυρία Γκρέσλε, και πάλι το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την συνεργασία. αυτό είναι το περιεχόμενο του, ε, κειμένου της κυρίας Γκρέσλε που θα το είχε αναγνώσει η ίδια, αλλά δεν πρόλαβε λόγω της ε, ψηφοφορίας μας. Με λίγα λόγια θα ήθελα τώρα να αναφερθώ σε, αυτόν τον κάπως περίπλοκο θεσμικό ελιγμό. Πρόκειται για τους απλοποιημένους δημοσιονομικούς κανονισμούς, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι να μπορέσει να υπάρξει άμεση απαλλαγή που δεν θα γίνει μέσα στα πλαίσια της Γενικής Απαλλαγής για την Κομισιόν μέσα από τον οικονομικό έλεγχο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και η Κομισιόν και περνώ στα αγγλικά αποφάσισε να αναθεωρήσει και υποσχέθηκε να αναθεωρήσει τον δημοσιονομικό κανονισμό στο προσεχές μέλλον. Μεταξύ των θεσμικών οργάνων μπορεί να γίνει μια προσπάθεια για την ε, χορήγηση άμεση απαλλαγής της μεγάλης DGI και θεωρώ ότι αυτό πρώτον εξασφαλίζει μια διαφάνεια, δεύτερον δίνει και μια άμεση απαλλαγή και στις συμμετέχουσες βιομηχανίες. Αυτό πρέπει να γίνει βέβαια με συνεργασία πολλών κοινοβουλευτικών επιτροπών και γι' αυτό ευχαριστώ ιδιαίτερα το Συμβούλιο το οποίο έδειξε κατανόηση και ε, συμμερίστηκε την προσπάθειά μας. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Η ελληνική προεδρία είναι παρούσα. Έχετε το λόγο. Η πρώτη σας ομιλία στην Επιτροπή μας. Thank you very much, Madam Chair. Indeed, it is our first uh, speech on the, the Parliament. Thank you very much. Πράγματι είναι η πρώτη μας ομιλία στην Επιτροπή σας να ενημερώσω ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης Πάρτε 1 που έγινε χθε, καταλήξαμε σε μια συνενετική δήλωση για μια ξεχωριστή απαλλαγή για τα joint undertakings. Η Προεδρία κατέληξε ότι η κοινή δήλωση θα δοθεί στο Συμβούλιο προς έγκριση. Σε αυτό το πλαίσιο περιμένουμε μια επικοδομητική αντίδραση από πλευρά σας έτσι ώστε να προχωρήσουμε με το πακέτο καινοτομίας σημαντικό ε, και θεωρούμενο κατά προτεραιότητα θέμα. Ευχαριστώ πολύ Κομισιόν. Ευχαριστούμε. Καλό, καλή χρονιά πρώτα απ' όλα. Χαιρόμαστε γιατί επετεύχθη αυτός ο συμβιβασμός. Αυτό καταδεικνύει την καλή συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων, το οποίο είναι και εχέγγυο βεβαίως επιτυχίας. Ε, ε, πρέπει να πούμε ότι αυτό το light financial regime μας ικανοποιεί, από την άλλη πλευρά βεβαίως. Χαιρόμαστε γιατί υπάρχει ε, μεγάλη διαφάνεια μέσω αυτής της απαλλαγής και αυτό μας ε, ευχαριστεί κυρίως γιατί αποτελεί και επιστέγασμα των προσπαθειών που κάναμε έτσι ώστε να προωθήσουμε το θέμα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Η συνάδελφος Σόγερ Μαντουρέλ. Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να πω εξ ονόματος της πολιτικής μου ομάδας ότι καλωσορίζουμε την ελληνική προεδρία εμείς εκφράζουμε την ευαρέσκειά μας και για τη συμβιβαστική λύση στην οποία καταλήξαμε. Αυτή ήταν η πρότασή μας εδώ και καιρό. Ελπίζουμε να προχωρήσει η συμφωνία αυτή και να εφαρμοστεί το ταχύτερο δυνατόν. Κάτι το οποίο θα είναι χρήσιμο και για το θέμα της, ε, του, του του ορίζοντος 2020 Νομίζω ότι ε, δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω στην παρούσα φάση. Ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχει άλλο εγγεγραμμένος ε, ομιλητή και επομένω, ε, εάν δεν ζητά κάποιος άλλος το λόγο μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Α, κύριε Έλλερ, θέλετε το λόγο, παρακαλώ. Ο κύριος Έλερ, πάλι, μία παράκληση αγγλικά. Το συζητήσαμε ήδη στην πρώτη συνάντηση των σκιωδών εισηγητών και επειδή πρόκειται από τα πιο σημαντικά οριζόντια θέματα, θέλω να βεβαιωθώ ότι όλες οι πολιτικές ομάδες έχουν την ίδια γνώμη, διότι έχουν κατατεθεί διάφορες τροπολογίες, αλλά μία καταρχήν, μία κατά οριζόντια τροπολογία, με την οποία συμφώνησαν οι ε, σκιώδεις εισηγητές, αλλά επειδή δεν έχει υπάρξει ρητή αντίδραση άλλων πολιτικών ομάδων. Την ε, γνώμη αυτή μοιράζονται μεν Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και Σοσιαλδημοκράτε, αλλά θα ήθελα να γνωρίζω εάν την άποψη τη ίδια απόψη μοιράζονται και οι άλλε πολιτικέ ομάδε που είναι παρούσε εδώ. Βλέπω κάποιου να ανέβουν καταφατικά. Καλά, αυτό ήθελα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, θέλετε το λόγο. Παρακαλώ, συνάδελφε. Λοιπόν, ζήτησα το λόγο για να ρωτήσω το εξής. Ε, αυτή η συμφωνία ε, περιλαμβάνει και θέματα όπως ε, μείωση του προϋπολογισμού και άλλα θέματα τα οποία συζητήσαμε. βλέπω τον κύριο Έλληρο ότι νεύει αρνητικά, επομένως ναι, ναι, μιλάμε μόνο για την απαλλαγή, επομένως δεν υπάρχει πρόβλημα. Πρόεδρος, έχει το λόγο για κύριο Βανίστεροι. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ λοιπόν με αυτά που υπόθηκαν. Όλα αυτά είναι πολύ ευαίσθητα θέματα. Ε, ε, πρέπει βεβαίως ε, να γίνεται διαπραγμάτευση από την άλλη πλευρά. δεν πρέπει να αποτελματώνεται η συζήτηση. Πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσουμε να προχωράμε τις διαδικασίες έτσι ώστε να υλοποιούνται και τα προγράμματα. Θα πρέπει να ξεπεράσουμε γρήγορα και όλα αυτά τα δημοσιονομικά ζητήματα. Η μόνη ε, προσέγγιση που ε, ε, είναι ικανοποιητική είναι η δουλειά η οποία ολοκληρώνεται. Γιατί έχουμε πίεση όσον αφορά τα οικονομικά ζητήματα. Απ' την άλλη πλευρά ε, πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε κατά νου τους ε, κύριους στόχους και όχι μόνο να κόβουμε από το ένα πρόγραμμα για να δίνουμε στο άλλο και να ανακυκλώνουμε τα χρήματα. Αυτό το έχουμε συζητήσει επανειλημμένα με τους σκιώδεις. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί. Πρόεδρος, δεν έχω κανένα εγγεγραμμένο αγορητή, λέει η Πρόεδρος πλέον και επομένως δεν ξέρω αν θέλει η Κομισιόν να προσθέσει κάτι. Όχι. Ούτε η Προεδρία από ό,τι βλέπω. Επομένως, μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτήν την πολύ πυκνή πρωινή συνεδρία. Η ψηφοφορία στην Ήτρε θα γίνει την 5η 24 Ιανουαρίου και η συνεδρίασή μας θα λάβει χώρα 22 και 23 ε, Ιανουαρίου στις Βρυξέλλες. Ε, ε, κύριε Έλερ. Ζητώ συγγνώμη, ε, δεν θέλω να καθυστερήσω, αλλά παρόλα αυτό να ζητήσω από τους συναδέλφους ε, να είναι παρόντες στην επόμενη συνάντηση των σκιωδών εισηγητών. Όπως είπε και ο κύριος Βανίστερόι, ε, έχουμε πολλά να συζητήσουμε για τον προϋπολογισμό και για άλλα παρεμφερή θέματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προχωρήσει η συμφωνία με το Συμβούλιο ε, πρέπει να δούμε και τι κάνουν οι συνάδελφοι στην Επιτροπή Κοντ ε, και να δούμε και κάποια οριζόντια ζητήματα τα οποία αφορούν ε, σειρά εκθέσεων. Επομένως, η επόμενη συνάντηση των σκιωδών εισηγητών είναι θεμελιώδου σημασίας. Παρακαλώ και καλώ όλους τους συναδέλφους σκιώδης εισηγητές να είναι παρόντες. Συνεχίζει χωρίς μικρόφωνο ο κύριος Έλερ, δεν ακούν οι η κυρία Μαζίτ Κόμψ είχε ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι χρειάζεται να γίνει η συνάντηση των σκιωδών την επόμενη εβδομάδα. Ελπίζω να είναι εφικτή η σύγκληση αυτή. Είμαι σκιώδης επίσης και για το πρόγραμμα Eurostar. Το πρόγραμμα Eurostar είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις λεγόμενες startups, τις μικρές επιχειρήσεις που ξεκινούν τη δραστηριότητά τους. Μιας και έχουμε τη συμβιβαστική πρόταση, ε, θα πρέπει να τη συζητήσουμε, γιατί δεν έχουμε συζητήσει για τη συμβιβαστική αυτή πρόταση. Είναι τόσο σημαντικό το θέμα αυτό, που θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε σήμερα, αλλά τώρα πια δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Απλά θα ήθελα να υπογραμμίσουμε ακόμα περισσότερο το θέμα αυτό, γιατί θα βοηθήσει τις ε, ε, επιχειρήσεις που ξεκινούν τώρα. Κοιτάξτε, είχαμε μια πολύ δύσκολη μέρα, λέει η κυρία Σαρτόρη, και γι' αυτό η συζήτηση και αυτή είναι λίγο περίεργη. Η κυρία Καρβάλιο έχει το λόγο. Μια διευκρίνηση έγιναν κάποιες συζητήσεις τις οποίες δεν προσεκλήθη γιατί νόμιζα ότι είναι μόνο για τους εισηγητές και όχι για τους σκιώδεις. Παρακαλώ αν οι συναντήσεις αυτές περιλαμβάνουν και τους σκιώδεις πρέπει να αποσταλούν και σε αυτούς προσκλήσεις. Προς το παρόν εγώ δεν έχω κληθεί σε καμία από τέτοιες συναντήσεις. Ξέρω ότι γίνονται συναντήσεις ανάμεσα στους εισηγητές αλλά δεν έχω λάβει προσκλήση, πρόσκληση ε, ως ε, σκιώδη εισηγήτρια. Θα πρέπει λοιπόν να σταλούν προσκλήσεις και στους σκιώδεις. Η Ριέρα Μαντουρέλ. Να διευκρινίσω λίγο το συγκεκριμένο θέμα. Εμείς εργαζόμαστε ε, ξεχωριστά ο κάθε ένας εισηγητής βέβαια και συνεργαζόμαστε ο καθένας με τον σκιώδη του, με τους σκιώδεις που ασχολούνται με τη συγκεκριμένη έκθεση και συνεργάζονται και μεταξύ τους ε, οι εισηγητές. Εγώ δεν θα είχα κανένα πρόβλημα αν θέλετε στις συναντήσεις αυτές να προσκαλούνται και οι σκιώδεις, ίσως να γίνει πιο αποτελεσματική. Για τις τεχνικές συναντήσεις αύριο σαν παράδειγμα υπάρχει μια οριζόντια τεχνική συνάντηση ε, γύρω από όλα τα θέματα αυτά έτσι ώστε να υπάρξει καλύτερο συντονισμός. Τεχνική συνάντηση. Η αυριανή είναι μια τεχνική συνάντηση, επαναλαμβάνω. Στην περίπτωσή μου, σαν παράδειγμα, στην περίπτωση του Ήμι την Δευτέρα, έχω μια συνάντηση με όλους, τις, με όλους τους σκιώδεις της Επιτροπής. Προβλέπονται τέτοιου είδους συναντήσεις λοιπόν των εισηγητών και μπορούμε να προσκαλέσουμε και τους σκιώδεις. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Απλά εξήγησα τη διαδικασία μέχρι σήμερα. Κοιτάξτε είναι σαφές τώρα πια λέει η κυρία Καρβάλιο ότι δεν έχουν προϋπάρξει συναντήσεις και με τους σκιώδεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Uh, το θέμα αυτό για μένα ήταν σημαντικό. Το θέμα είναι να βελτιώσουμε τις δυνατότητες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι σημαντικό τμήμα των θέσεων απασχόλησης, μεν, αλλά στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης έχουν μόνο το, αντιπροσωπεύουν μόνο το 4%. Αυτό το 4% λοιπόν στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης ε, και ε, το 70% που είναι ε, το ποσοστό δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης είναι κάτι το οποίο πρέπει να γεφυρώσουμε με τη βοήθεια και των ευρωπαϊκών μέσων, οργάνων αν θέλετε. Η διαπραγμάτευση αυτή λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι κάτι το οποίο βοηθά να ξεπεράσουμε τις διαφορές ανάμεσα στις χώρες Υπάρχουν σημαντικές εμπειρίες στις βόρειες κυρίως χώρες. Ξέρετε ότι στη Δανία υπάρχουν ε, πολύ μικρές επιχειρήσεις κάτω των 10 υπαλλήλων που μπορούν παρόλα αυτά να λειτουργήσουν με εξωστρέφεια σε διεθνές επίπεδο. Η πρωτοβουλία αυτή λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία και θα συνεισφέρει στην αναζωογόνηση νομίζω των ευρωπαϊκών οικονομιών. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας εμείς έχουμε προετοιμάσει εννέα συμβιβαστικές ε, προτάσεις. Έχουμε φέρει κοντά τις θέσεις μας ο ένας τον άλλο και θεωρώ ότι η συνάντηση των σκιωδών ε, στην παρούσα φάση δεν είναι ε, απαραίτητη γιατί μπορούμε να επικοινωνούμε με ηλεκτρονικό τρόπο πολύ εύκολα και αρνούμε την πρόταση του κυρίου Έλερ να μειώσουμε δηλαδή ε, τις πιστώσεις κατά 12,5% είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να δεχθώ σε καμία περίπτωση. Γιατί αυτό θα σταματήσει ουσιαστικά κάθε πρόοδο στον συγκεκριμένο τομέα. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Έλερ έχει το λόγο. Θα δώσω το λόγο και στην κυρία Ματζέη Κούκοβιτς πρώτα και μετά θα κλείσουμε. Να εξηγήσω τη διαδικασία, επιμένει ο κύριος Έλερ. Ο λόγος για τον οποίο συναντήθηκαν οι συγητές και σκιώδεις συγητές είναι ότι προσπαθήσαμε να φτιάξουμε μια ατζέντα για το οριζόντιο θέμα, την οριζόντια τροπολογία. Δεν έχει ε, νόημα να υπάρχουν διαφορές ε, για τις διάφορες κοινέ επιχειρήσεις. Θα πρέπει να υπάρχουν οι ίδιες, οι ίδιοι κανόνες και η ίδια διάρκεια για τις απαλλαγές. Γι' αυτό συναντήθηκαν οι εισηγητές. Και εγώ θα ζητούσα να μην κατακαιρματιστούν όλες αυτές οι εκθέσεις και να προτείνουν διαφορετικές λύσεις γιατί κάτι τέτοιο δεν θα αποδώσει. Γι' αυτό και συναντηθήκαμε πριν από τα Χριστούγεννα. Το δεύτερο θέμα είναι ότι κάθε επιμέρους εισηγητής καλείται τώρα να συναντηθεί με τους κοιόδης να του ζητήσει να συμφωνήσουν με την έκθεσή του, έχοντας ταυτόχρονα υπόψη ότι εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη για μια οριζόντια συμφωνία. Σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό, εγώ πρότεινα ένα αριθμό, ένα νούμερο για τον προϋπολογισμό, έχοντας υπόψη ότι δεν είναι cherry picking, έχουμε 16% περικοπή του προϋπολογισμού. Είτε θα απηχείται αυτό και επομένως θα είναι ίδιες περικοπές σε όλα τα προγράμματα, ή περικόπτουμε όλα τα προγράμματα εκεί όπου είναι και περικόπτουμε περισσότερο GDIs και PPPs. Εν τέλει νομίζω θα είναι σκόπιμο να υπάρξει μια, ε, ένας οριζόντιος συμβασμός στον προϋπολογισμό μπορεί με ίσως διαφορετικές μεμονωμένες προτάσεις αλλά δεν έχει νόημα να έχουμε μια συνολική περικοπή και αυτή να μην έχει απήχηση στον προπολογισμό, διότι η περικοπή υπάρχει, δεν μπορούμε να την αποφύγουμε. Νομίζω ότι θα πρέπει να επιδιώξουμε να ορίσουμε όπως το κάναμε τα οριζόντια θέματα και μετά να ψηφίσουμε κάτι περικοπή όχι, αλλά κάπως πρέπει να βγει πολιτικά, διότι γίνεται ο περικοπή στο προπολογισμό και αν δεν το κάνετε εκεί θα πρέπει να βγει κάπου αλλού. Γι' αυτό άλλωστε όπως είπα συναντήθηκαν οι εισηγητές. αλλά δεν είναι η τελική λύση αυτή. Λαμβάνουμε τώρα τις τροπολογίες, θα επιδιώξουμε να καταλήξουμε σε συμβαστικές τροπολογίες και αυτή είναι η δουλειά εισηγητών και σχεδόν εισηγητών, αλλά θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία μεταξύ των πολιτικών ομάδων για το οριζόντιο θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, συζητάμε λίγο άτυπα τώρα πλέον, κυρία Ματέη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ θα ήθελα να πω ότι μέσω του προγράμματος Eurostar στην ουσία συζητάμε για 10.000 θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργηθεί στο παρελθόν και στο μέλλον θα δημιουργηθούν ακόμα περισσότερο μέχρι το 2020. Ε, ακριβώς λόγω αυτού πρέπει να δείξουμε ε, υπευθυνότητα οι συγητρίες και οι συγητές ε, θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον μία συνεδρίαση. Δεν είναι δυνατόν να πούμε ότι μπορούμε να τα λύσουμε όλα μέσω ηλεκτρονικής συνεννόησης. Μιλάμε εδώ για τις ζωές των ανθρώπων. Ε, μιλάμε για τη ζωή των ανθρώπων στο μέλλον, για το αν θα έχουν και τι είδους εργασία θα έχουν, ποια θα είναι η απασχόλησή τους. Νομίζω ότι εμείς σαν Ευρωπαίοι βουλευτές θα έπρεπε οπωσδήποτε να βρούμε χρόνο για να συζητήσουμε για τέτοια πράγματα. Το email έχει την αξία του, αλλά δεν πάβει να είναι ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Άλλο είναι η ζωντανή συζήτηση. Ευχαριστώ κύριο Σοντή. Ο κύριος Σοντή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστούμε και τον συνάδελφο ε, Κρίστιαν Έλερ, ο οποίος με μεγάλη υπομονή συντονίζει όλα τα θέματα αυτά. Έχω να κάνω πολλές παρατηρήσεις. Πρώτον, επίγει η κατάσταση σε σχέση με την υλοποίηση, γιατί αυτές οι ε, κοινέ ε, επιχειρήσεις περιμένουν τα κείμενα. Είναι κείμενα τα οποία στην ουσία είναι υποπροϊόντα του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Ε, εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, δεν πρόκειται να ανατρέψουμε όλες τις καταστάσεις μέσα σε ε, μερικές εβδομάδες πριν το τέλος της θητείας μας, αλλά παρόλα αυτά επίγει να αντιμετωπίσουμε εγκάρσια και ε, ταχύτατα τα θέματα αυτά. Όσον αφορά τον προϋπολογισμό δεν θα περάσουμε ώρες επί ωρών να συζητάμε αν χρειάζονται 100.000 εκεί, ε, εκατομμύρια εκεί ή 100, εκατομμύρια εδώ. Εδώ ε, αναφερόμαστε σε, μια, σε ένα υπόδειγμα, σε ένα πρότυπο συνεργασίας ανάμεσα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Ας ολοκληρώσουμε τον προϋπολογισμό ε, με ενδεχομένως μία ε, γενική μείωση του προϋπολογισμού που όμως θα επιτρέπει την άμεση υλοποίηση των προγραμμάτων ας πάρουμε, ας καταλάβουμε ότι παίρνουμε πρόσκαιρες προσωρινές συζητήσεις διότι είχαμε την πρόνοια και τη Σοφία να περιλάβουμε και μία διάταξη στις ε, ε, αποφάσεις μας ε, μια διάταξη αναθεώρησης. Θα έχουμε επομένως την δυνατότητα να αναθεωρήσουμε του τους προϋπολογισμούς αυτών των κοινών επιχειρήσεων. Επαναλαμβάνω λοιπόν αυτό που είπα και στην αρχή. Εγκάρσια ταχύτατη αντιμετώπιση. Έχουμε μπροστά μας τις ευρωπαϊκές εκλογές, θα πρέπει να πούμε. Είμαστε υπέρ ή είμαστε κατά αυτών των κοινών επιχειρήσεων. Ε, και επαναλαμβάνω ότι στα πλαίσια της πολιτικής, της ρήτρας πολιτικής αναθεώρησης θα έχουμε τη δυνατότητα να αναθεωρήσουμε και προϋπολογισμούς και θέσεις κτλ. Αλλά Παρακαλώ πολύ εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προχωρήσουμε γρήγορα ε, διότι θα πρέπει ε, αυτά τα ε, κονδύλια να προχωρήσουν. Όσον αφορά τα κονδύλια για τον προπολογισμό θα τα αποφασίσει το επόμενο Κοινοβούλιο. Τελευταία παρέμβαση λέει η Πρόεδρος γιατί ούτως ή άλλως έχουμε φτάσει στις 12.30 και πρέπει να ολοκληρώσουμε η κυρία Ριαρ Μαντουρέλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να θυμίσω μετά από όλη αυτή τη διακοπή ότι το διάλειμμα αυτό είχαμε λοιπόν μια μεγάλη συνάντηση των σκιωδών όπου τέθηκαν και συζητήθηκαν όλα αυτά τα θέματα και τα οριζόντια και να συμφωνήσω με αυτά που είπε ο Σέλερ. Η πρόταση αυτή δεν είναι μια πρόταση η μείωση αυτή του κυρίου Έλερ. Είναι μια πρόταση η οποία επιβλήθηκε από τη γενικότερη μείωση του προϋπολογισμού στην οποία συμφώνησε και το Κοινοβούλιο. Πρόκειται για μια συνολικότερη μείωση την οποία πρότεινε το Συμβούλιο και δέχτηκε το Κοινοβούλιο για να καταλήξουμε σε μια γενικότερη λύση. Είναι σημαντική η μείωση αυτή, αλλά νομίζω ότι παρόλα αυτά είναι ελεγχόμενη και μπορούμε να την κατανείμουμε σε όλα τα προγράμματα που περιλαμβάνονται στον ορίζοντα 2020 και στις ε, κοινέ πρωτοβουλίες και Θα προσπαθήσουμε στο ίδιο ποσοστό λοιπόν να κάνουμε προτάσεις σε όλες τις δραστηριότητες που έχουμε μπροστά μας. Θέλω λοιπόν ότι εμείς σαν πολιτική ομάδα βέβαια συμφωνούμε με την πρόταση του κυρίου Έλλερ και να πω και στους άλλες, ήθελα απλά να θυμίσω στους συναδέλφους το ιστορικό της υπόθεσης αυτής. Βέβαια τα προγράμματα όπως το Eurostar έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και είναι θέματα τα οποία ίσως θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν και με διαφορετικό τρόπο. Πάντως να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα μιας ε, εξίσου μείωσης αν θέλετε και σε σχέση με τα GTIs και σε σχέση με τα υπόλοιπα προγράμματα. Αυτά είναι τα συμπεράσματα στα οποία είχαμε καταλήξει ε, στην πρώτη συνάντηση. Πάντως αυτή είναι η γενική ιδέα και έτσι θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε τις συζητήσεις και να καταλήξουμε σε μια καλή κατανομή της μείωσης. Αυτή η συζήτηση έγινε στα πλαίσια της συνάντησης των σκιωδών ή των συνάντηση, ποια συνάντηση είναι αυτή που προηγήθηκε, επαναλαμβάνει η κυρία Καρβάλιο. Κοιτάξτε, έγινε στην οριζόντια συνάντηση όλων των εισηγητών, των εισηγητών, λέει η, η κυρία Μαντουρέλ. Καλώς διευκρινίστηκαν τα πάντα, λέει η κυρία Σαρτόρη, διακόπτουμε. Η ψηφοφορία προβλέπεται να γίνει στις 23 Ιανουαρίου. Καλή σας όρεξη.